μεταξύ των διαφόρων συστημάτων παραγωγής, εργασίας και μεταφορών. Και γι' αυτό θα ενεθάρρυνα τοπική και πράσινη παραγωγή. Ευχαριστώ. Μουτσουμέσκ, αγαπητοί συνάδελφοι Κούτας. Η κυρία Μπέρμπερ, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ.